να σας ενημερώσω για το εξή, για τις ε, δηλώσεις που έγιναν και δημοσιεύτηκαν βάσει το άρθρου 231 χθες στην ε, ε, Ολομέλεια. Δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις.